18 Ιουνίου για την εκλογή του κυρίου Μαουρίτσιο Έντζο Λούπι ως ε, Ευρωβουλευτού. Ωστόσο, μέχρι σήμερα ο κύριος Λούπι διατελεί υπουργό Μεταφορών και Υποδομών. Ε, πράγμα ασυμβίβαστο, σύμφωνα με το άρθρο 7 της πράξης 20 Σεπτεμβρίου 1976, ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτού, το να είσαι μέλος Υπουργικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 ε, του κανονισμού διαπιστώνει το Κοινοβούλιο όπως σήμερα τη χειρία της ε, παρούσης έδρας. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ακολουθεί εκλογή των αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω λάβει